Uh, good afternoon, colleagues, and thank you. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην συνεδρίασή σα στην αίθουσά σας για να κάνουμε αυτή την κοινή ανταλλαγή απόψεων για το πρόβλημα των αναγκαστικών εκτοπίσεων. Όπως ξέρετε, θα συντάξουμε από κοινού μια έκθεση για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα της κινητικότητας προσφύγων και μεταναστών. Είναι θέμα προτεραιότητας τη σημερινή μέρα και όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, ε, μια λύση ανθρώπινη για όλους αυτούς τους ανθρώπους αλλά θα πρέπει να είναι βέβαια και βιώσιμη η λύση και να μπορούσουμε να υποδεχθούμε τους ε, ανθρώπους αυτούς και άπαξ και εκτοπίζονται τουλάχιστον να την χάνουν καλής μεταχείρισης. Και επίσης στις 19 Σεπτεμβρίου έχουμε μια διάσκεψη του ΟΗΕΠ όπου θα, θα ζητηθούν αυτά τα ζητήματα. μεταξύ των οποίων δηλαδή θα ζητηθεί και η εκτόπιση. Έχουμε τώρα ως βάση συζήτηση την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχει εγκριθεί το κείμενο και από το Συμβούλιο. Έχουμε επομένως τρει τρεις καλεσμένους. Έχουμε τον κύριο Ντεμπράουερ από την ΕΚΟ, τον κύριο Αμπρόζη από την Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης και είναι η κυρία Χάλντ από το Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Κύριε Ντεμπράβο, αν θέλετε πέστε μας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επειδή αργήσαμε να ξεκινήσουμε και επειδή έχω κάποια άλλη υποχρέωση θα πρέπει να σας εγκαταλείψω πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Λέει η κυρία Μάκαβαν. Ωραία, ωραία, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Πρόεδρε. Ξέρω, ξέρω ότι είμαστε πίσω στο χρονοδιάγραμμα, οπότε και θα περιορίσω αυτά που θα σας πω στα βασικά του μηνύματος, μια που έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Αυτή δημοσιοποιήθηκε εδώ και πολύ καιρό και πέρασε και εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο, όπως μας είπατε, κυρία Πρόεδρε. Και επομένως τα βασικά σημεία του κειμένου είναι γνωστά. Οπότε ε, να ξεκινήσω εγώ, να τα πούμε μετά οι άλλοι συνάδελφοι εδώ και θα έχουμε εδώ τα απαντήσει μετά. Είπαμε ότι εδώ είναι ένα ολόκληρο μοσαϊκό. Αυτό είναι μόνο μια ψηφίδα. Έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε το, θέμα του πώς θα το διαχειριστούμε ε, και έχουμε το πρόγραμμα δράσης. Ε, αυτά είναι τα θεματολόγια και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε και να πάμε έτσι στο, στη συνάντηση κορυφής για την ανθρωπιστική μας πολιτική. Οπότε ακριβώς στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο θα γίνει συνάντηση που προείπαμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τώρα, τι, τι, στοχεύει αυτή η ανακοίνωση να τα ξαναθυμηθούμε τα βασικά σημεία. Ότι έχουμε 65 εκατομμύρια ε, των εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο. Είναι ρεκόρ αυτό στο οποίο φτάσαμε. Αλλά επίσης ε, πέραν αυτών είπαμε ότι έχουμε εκτοπίσεις από Σομαλία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν ε, και έχουμε επίσης τρεις από τους βασικότερους πέντε σε όλο τον κόσμο, Συρία, Κολομβία, Σουδάν. Αλλά γιατί έχουμε την παράταση αυτής της εκτοπής πάνω από τα πέντε χρόνια, γιατί έχουμε τέτοιου είδους εκτοπισμό και εσωτερικό εκτοπισμό, γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Πρόκειται για κάποιους που είναι ευάλωτοι, κάποιοι που υφίστανται τον, τον εκτοπισμό. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε πολλές κατευθύνσεις, γιατί συνήθως όλα θα γίνονται σε χώρες που ήδη χαρτίζονται από κάποια ευπάθεια, ήδη άνθρωποι και είναι ευάλωτοι. Είναι περιοχές όπως η Αιθιοπία, όπως το Σαχέλ, όπου σοβούν κρίσεις. Άρα ο εκτοπισμός είναι αποτέλεσμα περιπλόκων καταστάσεων. Και βλέπουμε ότι το ένα πρόβλημα δημιουργεί το άλλο. Άρα εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε στο για ποιους λόγους είναι ευπαθείς αυτές οι ομάδες ανθρώπων. Και βεβαίω και θα αναλυθεί αυτό και από τους ε, παρακαθημένους μου, τι γίνεται με τα τι γίνεται με τους ε, πρόσφυγες, από πού προέρχονται, αλλά δεν είναι αυτό το δικό μας θέμα. Το δικό μας θέμα είναι το πώς θα καλύψουμε το πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μετανάστες. Ε, γιατί ακριβώς γίνονται ευάλωτοι μια που μετακινούνται και γιατί παρατείνεται ε, αυτή τους η κατάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Ε, αυτό είναι φαινόμενο που προϋπήρχε πριν εγώ ασχοληθώ με το θέμα στην Κομισιόν στη Λατινική Αμερική και στην Ασία, παλαιότερα μετά στην Αφρική. Οπότε αυτή η παρατεταμένη εκτόπιση είναι κάτι το παλιό. Άρα για να κάτσουμε να δούμε το έγγραφο εργασία που προσαρτάται στην ανακοίνωσή μα, θα δείτε ότι έχουν γίνει πολλέ προσπάθειε στο παρελθόν, τόσο ώστε να υπάρχει προσέγγιση με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στην κάθε περίπτωση. Και συνήθω τι συμβαίνει, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια έρχεται πρώτη και επειδή πολλές φορές παρατείνεται η κατάσταση, ε, τότε ε, φτάνει στα ωριά της η ανθρωπιστική ενίσχυση για κάτι θα πρέπει να γίνει. Να, και τότε σκεφτήκαμε αυτό το LRRR, δηλαδή ε, βοήθεια, ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη. LRRD στα αγγλικά. Όμως το θέμα ήταν το τι πόροι υπάρχουν, τι οικονομικοί πόροι υπάρχουν γιατί το θέμα είναι ότι τελικά υπήρχε και η παγίδα της εξάρτησης. Δηλαδή αυτό το έχετε δει όταν πάτε στους καταβλισμούς, στα στρατόπεδα των εκτοπισμένων και των προσφύγων ότι κάποια στιγμή ε, το θέμα του ανθρωπισμού και της αξιοπρέπειας χάνεται, χάνεται αυτή η πτυχή γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι 100% από αυτή τη ρύθμιση και αυτό είναι το χειρότερο από όλα και πρόσφατα το διαπιστώσαμε επίσης μια που Τώρα έχουμε διάφορα σημεία όπου πηγαίνουν ε, οι Σύριοι στην Ελλάδα ας πούμε και περιμένουν όλη η μέρα να τους δώσουν ε, ένα πιάτο φαΐ να, γιατί μιλώ για ανθρωπισμό, για ανθρωπιά, για αξιοπρέπεια και σας παραπέμπω και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα της ε, Γενικής Συνέλευσης Άρα τελικά αυτό είναι το θέμα, η ανθρωπιά, η ανθρωπιστική μεταχείριση. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε για το πώς θα ασχοληθούμε πιο εμπειρικά. Θα αντιλήσουμε συμπεράσματα από το παρελθόν και πολλές φορές τα πήγαμε καλά, άλλες φορές δεν τα πήγαμε καλά. Ε, συντονισμός, επικοινωνία, πληροφόρηση, ε, ανεπαρκής πληροφόρηση, όλα αυτά έχουν συμβεί και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για τη νέα μας προσέγγιση. Άρα, για να δούμε, τι πρεσβεύουμε εμείς. Ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν υπάρχει παράταση αυτής της κατάστασης και πώς θα βρούμε κάποιες διαρκείς ε, λύσεις. Και πρέπει να δούμε τι, τι μας έρχεται, τι, έρχεται το στον ορίζοντα, τι υπάρχει και να έχουμε τους αντίστοιχους ε, πόρους για ανάπτυξη, για αρρωγή, ε, για ανθρωπιστική βοήθεια, να συνδέσουμε λοιπόν, την ανθρωπιστική βοήθεια με την ανάπτυξη και να γίνει τέτοια προσέγγιση, ούτω ώστε να προσπαθήσουμε ακριβώ όπω λέει και η ανακοίνωση από την εξάρτηση να πάμε στην ε, αυτάρκεια αλλά και παραπάνω. Δηλαδή αυτού του είδους η παρατεταμένη εκτόπιση ε, να ε, αποτελέσει εν σπέρματι μια ευκαιρία ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αναπτυχθούν για να γίνουν ε, κάποια εργονομένη κοινότητα. Αλλά βέβαια, να, ε, το καλύτερο παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται τώρα σε κάποιους καταβλισμούς στις Σομαλίας, μάλλον καταβλισμούς που πάνε Σομαλία εδώ και δεκαετία. Εκεί υπάρχει φοβερή εξάρτηση και δεν κατηγορώ κανέναν γιατί όλοι βάλαμε το δαχτυλάκι μας σε αυτή την κατάσταση. Και επαναλαμβάνω, μην με παρεξηγείτε γιατί βέβαια ασχολούμαι πολύ καιρό με το θέμα. Δεν κατηγορώ καμία πλευρά, αλλά κάποια στιγμή είχαμε ένταση μεταξύ της γύρω-γύρω κοινότητας και των ε, ε των εκτόπισμενο Ήταν μεγάλη ένταση. Και άρα θα πρέπει μακροπρόθεσμα να δούμε πώς θα έχουμε μια άλλη διαχείριση ε, του εκτοπισμού. Και πολλές φορές τι λέει η κυβέρνηση για διάφορους λόγους. Λέει ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση και παρεμβαίνει και δημιουργεί μια άλλη κρίση γιατί ακριβώς δεν υπήρξε διαχείριση που να λαμβάνει υπόψη το παρατεταμένο του εκτοπισμού εμείς όμως ξέρουμε τι πει παρατεταμένος εκτοπισμός και τι θα γίνει. Οπότε έτσι θα πρέπει να εμπλακούμε, έτσι θα πρέπει να ενισχύψουμε. Όμως πώς θα γίνει αυτό, γιατί ήδη έχουν πέσει διάφορες ιδέες. Να φέρει πίν. Το προηγούμενο πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας, το οποίο έγινε πρόγραμμα προστασίας και ανάπτυξης ευτυχώς για το κέρα της Αφρικής, αλλά και για τις χώρες Μαγκρέμπ Μασουρέκ ήταν ένα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε χέρι-χέρι με τους συναδέλφους της ανάπτυξης. Οπότε με τέτοια αντίληψη θέλουμε να προσπαθήσουμε αυτό το ψηφιδωτό να το συντεριάξουμε όσον αφορά την παρατεταμένη εκτόπιση. Τώρα όσον αφορά αυτά τα κατά πιστεύματα Ξέρω ότι έχετε πολλά ερωτηματικά για αυτά τα νέα μέσα και έχουμε και το Μαντάντ, το οποίο είναι λίγο υβριδικό, αλλά τέλος πάντων είπαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό το όργανο και έτσι να κάνουμε μια μόχλευση, μια από τον διάθεσή μας. Και έχουμε και άλλα προγράμματα διαμετακόμισης προς τη σωστή κατεύθυνση προγράμματα μεταφοράς, καμιά φορά ε, μπορούμε. Αλλά τι γίνεται με αυτούς τους οικονομικούς πόρους που θέλουμε να ε, ρίξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να τους κάνουμε υπεύθυνους αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί να καθορίσουν πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι που έχουμε διαθέσει να συμμετάσχουν στην τοπική οικονομία και να αγοράζουν εκεί από τους ντόπιου ό,τι χρειάζονται. Και έτσι βοηθάμε να αποκτήσουν και κάποια αξιοπρέπεια. Το έχω δει αυτό σε πολλά μέρη. Ξέρω ότι αυτό πολλές φορές θεωρείται μύθος, αλλά ε, υπάρχει, υπάρχει αυτό το θέμα. Από τη μια μεριά η ίδια η οικογένεια περιμένει να τους, να τους φέρουν πια φαΐ και οι υπόλοιποι του σπιτικού έχουν βγει να αγοράσουν από τους ντόπιου ε, χρήματα. Οπότε ε, αυτό τους δένει με τους ε, γείτονες, αλλά τους, ε, τους κάνει και καλύτερους. Οπότε, να, τι θέλουμε με αυτή την ανακοίνωση, να προωθήσουμε μία νέα προσέγγιση για την παρατεταμένη εκτόπιση. βεβαίω θέλουμε βιώσιμη λύση αλλά αυτά τα 65 εκατομμύρια που σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν αφορούν το 15 και αφορούν την μετεγκατάσταση γιατί έχουμε όλο ένα και περισσότερες εκτοπίσεις αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι έχουμε όλο ένα και λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ θα βάλω τελεία κυρία Πρόεδρε και θα δώσω τη σκητάλη στους ε, συναδέλφους, τους άλλους εμπειρογνώμονες και εκείνοι θα σας πούν κάποια άλλη προσέγγιση, ίσως που να μοιάζει με τη δική μου. Πάντως, είναι πάρα πολύ θετικό ότι έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και όπως σας είπα στην αρχή της εισήγησής μου, τώρα πρόκειται για ένα ευρύτερο θεματολόγιο το οποίο σχηματίζεται με επίκεντρο το μεταναστευτικό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά που έχουμε ήδη ε, πετύχει και στην συνάντηση του Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι για τον, ε, για τον... Ευχαριστούμε πολύ. Η ανάπτυξη με την ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι που ζητάνε συνάδελφοι εδώ και πολύ καιρό να το συνδυάσουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παντζέρη τώρα. Για να λάβετε την Προεδρία, αλλά πρώτον να δώσω το λόγο στην Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι γενικό διευθυντή, Μόνο διευθυντή είμαι. Τι να κάνω. Αλλά ποιο ξέρει, μπορεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να συμμετάσχω στην συζήτηση για ένα ζήτημα που βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό και που μας απασχολεί και μας πολύ και που βέβαια μας βάζει σε συνεργασία με άλλους φορείς, άλλους παράγοντες και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τελευταίο και το πρώτο τελευταίο σημείο που ανέφερε ο συνάδελφος, ότι η σύνδεση αυτή της ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανάπτυξη για να ανταποκριθούμε στην μεταναστευτική προσφυγική κρίση κλπ. είναι ένα κομματάκι μιας πιο συνολικής απάντησης που πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα. Ένα θετικό έχει βγει από την πρόσφατη αύξηση των μεταναστευτικών ουρών προς την Ευρώπη. Και αυτό είναι ότι αυτό που διαπιστώνουμε δεν είναι μια κατάσταση συγκυριακή, είναι συστημική, είναι διαρθρωτικό το ζήτημα και απαιτεί μια συστημική και διαρθρωτική απάντηση και όχι απλώς και μόνο μια συγκυριακή. Να δώσουμε δηλαδή μια απάντηση σε ένα επίγον ζήτημα που έχει προκύψει. Το θέμα που υπογράμμισε ο Σανλουίνε έχει να κάνει και με το εξή, ότι πρέπει να δούμε το πλαίσιο και άλλων ανακοινώσεων, πολιτικών και που έχουν προκύψει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους μήνες. Και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης και το πώς αντιμετωπίζουμε τη μετατόπιση των πληθυσμών των Ιούνιου. Για παράδειγμα, είχαμε κάτι για εταιρική σχέση όσον αφορά το μεταναστευτικό με τρίτες χώρες. Για μας, λοιπόν, Αυτά που συζητάμε έχουν να κάνουν με την προσπάθεια και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από τις χώρες μέλη και τη διεθνή κοινότητα γενικά για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της μετανάστευσης και άρα της μετατόπισης πληθυσμών. Και αυτό είναι ζωτική σημασία προκειμένου να δώσουμε μια απάντηση, να βελτιώσουμε την διαχείριση όχι μόνο της κρίσης, αλλά και της μετατόπισης πληθυσμών. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα, και όχι μόνο στην Ευρώπη, κυρίως όμως στην Ευρώπη, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι έχουμε μια ποικιλία, διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων που μας φτάνουν. Έχουμε την κλασική περίπτωση προσφύγων που έρχονται από περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε σύγκρουση και βέβαια χρειάζονται την προστασία μας. Έχουμε τους λαθροδιακινητές, δηλαδή τους ανθρώπους που περνάνε λαθροδιακινητές. Έχουμε αυτούς που μας έρχονται γιατί ψάχνουν καλύτερες συνθήκες ζωής, η εργασία, η εκπαίδευση μερικές φορές. Έχουμε συνεπώς ένα μείγμα ρόν ανθρώπων που φτάνουν δηλαδή στην ε, Ευρώπη και όλο και περισσότεροι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και όχι μόνο στην Ευρώπη και αλλού. Γι' αυτό λοιπόν και η προσέγγιση του να επικεντρωθούμε πρώτα απ' όλα στο πόσο ευάλωτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ βασικό. Να μην ασχοληθούμε δηλαδή μόνο με συγκεκριμένες κατηγορίες μην τους βάζουμε ταμπέλες και τους κατηγοριοποιούμε. Γιατί μπορεί κάποιος να μην φεύγει από μία εμπόλεμη ζώνη, παρόλα αυτά να πρέπει να το προσέξουμε ακόμα περισσότερο επειδή κινδυνεύει εξαιτία άλλων χαρακτηριστικών του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στο πόσο ευάλωτο είναι ένα άτομο που έρχεται στις χώρες μας. Να πω τώρα και δύο λόγια για κάποιες άλλες πτυχές, οι οποίες υπογραμμίστηκαν και στην προηγούμενη παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε, προσφυγική και μεταναστευτική κυρίως, Είναι μια παρατεταμένη κρίση. Άρα ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η παρατεταμένη κρίση θα έχει επιπτώσεις και στην εξέλιξη της κρίσης αυτής, στην εξέλιξη, σε εξελίξεις στη χώρα προέλευσης των ανθρώπων αυτών και στο ίδιο το μέλλον των χωρών από τις οποίες προέρχονται αυτοί. Σομαλία, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχει μια συνεχιζόμενη από το 92 ουσιαστικά, 24 χρόνια τώρα έχουμε τέτοια ε, κρίση εκεί. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν ως ε, πρόσφυγες όλη τους τη ζωή. Δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε εδώ μια ολόκληρη γενιά προσφύγων. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό για το μέλλον τους και για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη δικιά τους τη ζωή και τη ζωή των χωρών τους. Εξαιτία ε, λοιπόν της φύσης, της κρίσης που είναι παρατεταμένη, δεν πρόκειται για την εξαίρεση αλλά για τον κανόνα. Και γι' αυτό ακριβώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας με διαφορετικό τρόπο ευθύ εξ αρχής. Πρέπει να είμαστε σε θέση από την αρχή να δούμε ποια είναι τα πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα που προκύπτουν κάθε φορά που προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε, αναπτυξιακή βοήθεια, αντοχή, ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Να λάβουμε υπόψη μας από την αρχή δηλαδή το ότι πρόκειται για κάτι μακροπρόθεσμο και όχι κάτι που θα λήξει πολύ γρήγορα. Επίσης, πάλι επειδή κρατάει τόσο πολύ αυτή η κρίση, δεν πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν ε, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε μια χώρα, τους παρκάρουμε σε ένα καταβλισμό ή δεν ξέρω τι σε ένα χώρο που τους έχουμε προετοιμάσει περιμένοντας καλύτερες στιγμές για να επιστρέψουν στις χώρες τους. Γιατί ο χώρος αυτός που τους έχουμε παρκάρει, για να το πω έτσι, μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Χρειάζονται και ανθρωπιστικά μέσα και βοήθεια, αλλά και αναπτυξιακή βοήθεια ευθύ εξ αρχής, ώστε να βοηθήσουμε να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση και στις κοινότητες που φιλοξεχνούν τους ε, πρόσφυγες αυτούς. Να αποφύγουμε κοινωνικές εντάσεις που μπορεί να προκύψουν και που άρα θα δημιουργήσουν άρα επιπλέον προβλήματα στη διεθνή κοινότητα δευτερογενείς μετακινήσεις, υποβάθμιση του περιβάλλοντος γύρω από μεγάλους καταβλισμούς που έχουμε στον κόσμο, αλλά και άλλες τέτοιες καταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν για να σας πω ότι πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει με την ανακοίνωση αυτή και με άλλες και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών είναι ευπρόσδεκτες εξελίξεις κατά τη γνώμη μας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τα κατάλληλα εργαλεία και πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά και ότι θα ενισχύσουμε την ικανότητά μας να φέρουμε αποτελέσματα. Και βέβαια είναι και ένας προβληματισμός χωρίς τέλος, έτσι, η ανακοίνωση αυτή. Εννοείται ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ένα διαρθρωτικό ζήτημα, αλλά και ένα ζήτημα που διαφοροποιείται, αλλάζει με πολύ ταχύς ρυθμούς. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σε θέση να ανταποκρινόμαστε ανα πάσα στιγμή με την ίδια ταχύτητα. Θα σταματήσω εδώ με τα σχόλιά μου επί του θέματος και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε ή να συμμετάσχω, εν πάση περιπτώσει, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την άποψη του Συμβουλίου για τους πρόσφυγες της Δανίας σε σχέση με τη μετα... μετακίνηση και την ανάπτυξη θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες σκέψεις μου για την μεικτή μετανάστευση και την ανάγκη να σχεδιάσουμε καλύτερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από μια σύγκρουση και τις μακροχρόνιες λύσεις. Και θα επαναλάβω σε κάποιο βαθμό αυτά που είπαν οι δύο προλαλήσαντες. Οπότε δεν θα ακούσετε πολύ διαφορετικά πράγματα ίσως. Η παγκόσμια ανθρωπιστική διάσκεψη είναι το πρώτο θέμα που θέλω να αναφέρω. Ένα από τα πιο θετικά αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης ήταν η γενική αναγνώριση ότι η προσφυγική κρίση και η ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή θα είναι παρατεταμένη και αυτό απαιτεί μια μακροχρόνια απάντηση και πολιετή οικονομικό σχεδιασμό. Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ε, ανθρώπων που έχουν φύγει από τις αιστείες έχουν εκτοπιστεί για πάνω από 20 χρόνια. Το να βρούμε λοιπόν ε, μόνιμες λύσεις στις χώρες προέλευσης είναι απαραίτητο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε πολιτικές λύσεις σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις και παρατεταμένες συγκρούσεις. Το αναφέρατε και προηγουμένως ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πολιτικές λύσεις. Χωρίς πολιτι περισσότερη επένδυση στις πολιτικές λύσεις, ο αριθμός των εκτοπισμένων θα, συνεχίσει να αυξάνεται. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η α, παρατεταμένη κρίση σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις ε, ανθρώπινες ανάγκες και τις ανάγκες ε, προστασίας των ε, εκτοπισμένων που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης στις χώρες που είχαν υποδοχή, υποδοχής, όπως το τόνισε και η πρόεδρος της Επιτροπής σας που αποχώρησε, υπάρχει πάντα η πρόκληση της, ε, του παραδείγματος ανάπτυξης της χώρες όπου έρχονται οι εκτοπισμένοι. Τώρα με την αναγνώριση του παρατεταμένου χαρακτήρα θα πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη προγράμματος ανακουφιστικού χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να επανασχεδιάσουμε τις στρατηγικές ανάπτυξης για να λάβουμε υπόψη την μακροχρόνια διάσταση της εκτόπισης των ατόμων αυτών η κοινή αυτή συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Ανάπτυξης είναι και δείγμα το ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση του προβλήματος αυτού και θέληση να υπάρξει και διάλογος για τα θέματα αυτά. Μικτή μετανάστευση τώρα. Η μικτή μετανάστευση σημαίνει μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων, μεγάλη κλίμακος που είναι μετανάστες για διάφορους λόγους. Κάποιοι για τι χρειάζονται διεθνή προστασία και άλλοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι όλοι μια ομοιογενής ή αρμονική ομάδα και δεν έχουν όλοι δικαίωμα ασύλου, αλλά όλοι είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να τύχουν προστασίες. Νιώθουμε κάποια ανησυχία για τις πρόσφατες ε, Πρωτοβουλίε για την περιστολή τη μετανάστευσης στην Ευρώπη θεωρούμε ότι είναι κοντόφθαλμες και δεν θα περιορίσουν την πραγματική μετανάστευση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί ο αριθμό των μεταναστών που μπαίνουν στην Ευρώπη, αλλά φυσικά δεν μπορεί να μειωθεί ο αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται προστασία και δεν θα σταματήσει τις μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις δεν σταματάν, απλώς θα βρουν άλλους δρόμους για να φτάσουν στο στόχο τους αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό εμείς χαιρετίζουμε την έκκληση του Ban για να υπάρξει μια παγκόσμια συμφωνία για ασφαλή και τακτική μετανάστευση. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συμφωνία η οποία θα βασιστεί στις τωρινές ε, διμερείς και περιφερειακές ρυθμίσεις για τακτική και ασφαλή μετανάστευση και θα λάβει υπόψη τις ε, ευθύνες των χωρών προέλευσης, διέλευσης και, και, τελικού, και τελικού στόχου. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετανάστευσης με νόμιμο τρόπο που εξασφαλίζει την δυνατότητα ενσωμάτωσης των μεταναστών και καλύπτει και την ανάγκη ανθρωπιστικής απάντησης που θα εξασφαλίσει ότι η επιστροφή αυτών που δεν <clears throat> τηρούν τα διεθνή πρότυπα θα γίνει με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια καθώς και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίνοντας προτεραιότητα στην εθελοντική επιστροφή. Πρέπει να είναι μια συμφωνία που θα αναγνωρίσει τη θετική συμβολή των μεταναστών και των προσφύγων στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες υποδοχής και επίσης τη συμμετοχή τους στην εργασιακή δύναμη σε πολλές χώρες του κόσμου. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε μια συμφωνία η οποία μεταφράζεται σε συνεργασία επιτοπίως και σταματά την στεγανοποίηση η οποία δυσκολεύει τις απαντήσεις στις περιοχές όπου χρειάζεται πραγματικά συντονισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να, <clears throat> για να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια της μεταχείρισης όλων των μεταναστών επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και για να καταδείξει σε όλο τον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επομιστεί το τμήμα που της αντιστοιχεί για τις προσφυγικές ροές με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. ε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για τη μετανάστευση και γι' αυτό η τωρινή ρητορική για τους μετανάστες βασίζεται σε μεμονωμένες μοναχα και είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τη μετανάστευση, τι μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις και τι οδηγεί στην δευτερογενή μετανάστευση. Υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε την ικανότητα να αναλύουμε τα δεδομένα για τη μετανάστευση, ώστε να έχουμε συγκεκριμένα και αυτά στοιχεία τα οποία θα κατευθύνουν τις στρατηγικές μας. Μαζί με την ε, ύπατη ε, αρμοστία για την ε, μετανάστευση και την ούνρα, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη συλλογή στοιχείων για τη μετανάστευση. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε άλλες περιοχές όπως η Κεντρική Αφρική, η Δυτική Αφρική και η Κεντρική και Νότια Ασία πρώιμη σχεδίαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέρχονται από συγκρούσει. Αν ανατρέξουμε στην προηγούμενη εμπειρία από προηγούμενες σύγκρουσεις, ένα από τα κύρια διδάγματα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα πρώιμο στάδιο να αρχίσουμε να σχεδιάσουμε για μόνιμες λύσεις σε περιοχές συγκρούσεων. Παρά το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς πολλές φορές έχουν την ανάγκη να δώσουν μια άμεση βοήθεια, πρέπει να αναπτύξουν και σενάρια για μελλοντικέ βιώσιμες λύσεις. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων ατόμων και όπου δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς από τους πολιτικούς η μετατόπιση αυτή, εάν δεν γίνει σωστή σχεδίαση, η επαναφορά των ατόμων αυτών στις αιστείες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλοποίηση. Και οι βεβιασμένες ε, επιστροφές μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα. Η Κένια και Σομαλία είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Εάν δεν μπορέσουμε να μειώσουμε και να μετριάσουμε τους κινδύνους για την επιστροφή, όπως φάνηκε η Σομαλία, οι άνθρωποι αυτοί θα ξαναφύγουν. Μαζί με το Νορβηγικό Συμβούλιο και τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, το Δανικό Συμβούλιο για του πρόσφυγε προτείνει κοινέ πλατφόρμες στη Συρία με του εξή στόχου Να προωθήσουμε πρωτοβουλίε, οι οποίε μπορούν να υποστηρίξουν τη μελλοντική υποστήριξη στην ε, επιστροφή. Μπορεί να είναι προγράμματα νομική αρρωγή, όπω παραδείγματο χάρη στοιχεία πιστοποιητικά και τίτλοι ιδιοκτησία και δυνατότητε για οικονομική δραστηριότητα. Θα πρέπει να αναπτύξουν πλατφόρμες αυτές μια ανάλυση η οποία ενισχύει την υποστήριξή μας για το πώ η αλλαγή του πολιτικού χάρτη στη Συρία επηρεάζει τις ε, προοπτικές για τους πρόσφυγες, <clears throat> γιατί δημιουργείται ε, διαχωρισμός των πληθυσμών σε ομολογιακή και πολιτική βάση και πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες όλων αυτών των εκτοπισμένων ομάδων. Πολλοί από αυτοί δεν θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στις αιστείες τους ποτέ. Η πλατφόρμα αυτή πρέπει να οδηγήσει σε ένα σχέδιο λύσης το οποίο θα οδηγήσει σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε στοιχεία. Θα πρέπει να εντοπίσει τους κύριους παράγοντες των λύσεων που θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση για τη μελλοντική ε, επίλυση του προβλήματος των Σύριων προσφύγων και τέλος η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εμπλακούν στο να μεταλαμπαδεύσουν τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών που είναι εκτοπισμένοι για να υπάρξει η πρόκληση της καλύτερης λύσης και ασυγχρόνως έχουμε άλλη μια πρωτοβουλία στο κέρας της Αφρικής που είναι η <clears throat> ομάδα για την μόνιμη λύση που εργαστεί τα θέματα αυτά εδώ και δύο χρόνια. Τονίζουμε λοιπόν και την ανάγκη να ξαναβρούμε τα σωστά εργαλεία για την ανάπτυξη όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνιμες μορφές εκτόπισης, ζητούμε και μια, και μια παγκόσμια σύμβαση για τη μετανάστευση και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτά. Τρίτον, ενθαρρύνουμε περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της συλλογής δεδομένων και της καλύτερης διαχείρισης των πληροφοριών, ώστε να έχουμε μια πολιτική που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι απλώς σε αντίληψη της κατάστασης και για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε καλύτερα τι λύσει και τέλος ο σχεδιασμό για το μέλλον σε χώρε οι οποίες μαστίζονται από συγκρούσεις θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα και να συνάδει με τι προσπάθειε για την επίδευση πολιτικής λύση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμενους. Όλοι όσοι ήρθατε να αρχίσουμε τώρα τη συζήτησή μας, αλλά στις 6.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε τους δύο συνεισηγητές. Πρώτη είναι η Ελένα Βαλενσιάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τους ε, ειδικού μας. Μας εξήγησαν όλες αυτές τις ε, αρχές, ε, όλα αυτά τα οποία είναι θεμέλιο του προτινομένου συμφώνου. Εμείς θα πρέπει να αποπειραθούμε να συντάξουμε μία έκθεση που να παρουσιάζει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις και μας το είπανε καλύτερα πως εγώ μπορώ να το εκφράσω. Χρειάζεται ανθρωπιστική δράση, χρειάζεται πολιτική ανάπτυξη που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την ανθρωπιστική δράση. Άρα θα πρέπει όμως την έκθεση να δώσουμε και μια πολιτική διάσταση, δηλαδή την εξωτερική δράση. Και λόγω της τρομερής κρίσης των σύρων προσφύγων που, γιατί λέμε πρόσφυγες αφού τους απονείμαμε το καθεστώς που ήθελαν το καθεστώς του πρόσφυγα πρόκειται για κάποιους που ξέφυγαν, διέφυγαν, φυγάδες πολύ λίγοι από αυτούς χαρακτηρίστηκαν πρόσφυγες αλλά εμείς έτσι τους λέμε οι Σύροι πρόσφυγες άρα κοροϊδευόμαστε, παίζουμε με τις λέξεις τέλος πάντων, ακριβώς λόγω των ε, εκτοπισμένων σύρων συνειδητοποιήσαμε μέχρι ποιου σημείου αυτές οι εκτοπίσεις ανθρώπων τα επόμενα 20-30 χρόνια δεν θα σταματήσουν και μάλλον θα είναι φαινόμενο πιο γενικευμένο. Οπότε και θα πρόκειται για πολύ σημαντική πολιτική γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλές ε, πτυχές. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ε, ζητούν μια καλύτερη ζωή ή απλά να επιβιώσουν. Θα έχουμε επομένως τις αξίες μας. Θα έχουμε τους νόμους μας θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε το ότι άλλα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κάνει. Προτιωμένως για ανεξέλεγκτες μετακινήσεις κόσμου. Δεν υπάρχει κάποιο έφτακτη ασφαλής και αξιοπρεπής μετακίνηση. Ε, αυτό είναι πρόβλημα για την ασφάλεια και η ασφάλεια για τους πολιτικούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Ίσως οι περισσότερες αποφάσεις των τελευταίων μηνών σχετίζονται με την ασφάλεια. Οπότε και η ασφάλεια είναι κάτι που μας απασχολεί, γιατί αυτού του είδους μετακινήσεις των ε, πρόσωπων τούτων γίνονται και έτσι φουντώνει το αφήγημα των λαϊκιστών, των αντιευρωπαίων, των, των εξτρεμιστών, των ευρωφοβικών, οπότε θα πρέπει και εμείς να λάβουμε όπως για την πολιτική μας το πώς θα υπεραμεινθούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης της αλληλεγγύης ή όχι. Θα πρέπει, εν πάση αυτός ο προβληματισμός μας να αντιστοιχεί στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Και βεβαίως ε, όλα αυτά να συνάδουν με τις αξίες μας. Οι αξίες μας δεν αλλάζουν, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας. Και έτσι να βρούμε έναν συντονισμό καλύτερο, γιατί έχουμε πολλά μέτρα τα οποία δεν διέπονται από συντονισμό. Αυτό διαπιστώσαμε με όλους αυτούς τους ε, σύρους πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους πρόληψη της κρίσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φάση μετά τον πόλεμο, τη σύγκρουση. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στη, στην, τοπική πραγματικότητα για να μπορέσουμε να, να, να έχουμε ένα διάλογο με τις χώρες αυτές, που είτε από αυτές προέρχονται οι μετακινούμενοι, είτε είναι χώρες μέσα από τις οποίες περνάνε και να, προσπαθούμε να δώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση σε όλα αυτά. Χρειάζεται αλληλεγγύη και σεβασμός. Ακριβώς όπως είπαν και οι δικοί μας, άρα θα πρέπει και αυτό να σκεφτούμε για το πώς δηλαδή ε, θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς που μετακινούνται, που εκτοπίζονται. Φελή μπορεί να δουλέψει στο Βερολίνο και άλλος επειδή γεννήθηκε στον Νότο δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είπα ότι αυτό θα γίνει με μέτρα των Υπουργείων Εσωτερικών, αλλά θα γίνει και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα έτσι θα προχωρήσουμε στη σύνταξη του κειμένου, να δούμε πώς θα δώσουμε έναν τόνο κοινοβουλευτικό και εύστοχο για αυτή την προβληματική. Ευχαριστούμε. Αγκοστίν Διέθντε Μέρα τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Αντωνίου. Εκτιμάω ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις των προσκεκλημένων μας εδώ σήμερα το απόγευμα. Μας βοηθούν, μας βοηθούν στην εκπόνηση των εκθέσεών μας, και προκειμένου να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας. Τώρα, αυτό περί το οποίο πρόκειται εδώ είναι να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, τα θετικά που ακούσαμε σήμερα και να τα συμπεριλάβουμε στο έργο μας. Πιο συγκεκριμένα, για την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την ε, μετατόπιση πληθυσμών και της ανάπτυξης. Εμείς δεν είμαστε θεωρητικοί, είμαστε πολιτικοί, αλλά εμπειρικά γνωρίζουμε την τραγωδία αυτή και ιστορικά. Δεν είναι βέβαια τώρα η κατάλληλη στιγμή για να συζητάμε αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Η επαφή μας όμως είναι επαφή με μια τραγική πραγματικότητα επαφή με πρόσφυγες από ολόκληρο τον κόσμο σε μια πολύ σημαντική ιστορική στιγμή. Έχουμε να κάνουμε με μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμών τα τελευταία 30 χρόνια, κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι λοιπόν χρήσιμη αυτή η παρουσίαση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πρέπει να σας πω ότι από τη δικιά μου εμπειρία έχω διαπιστώσει ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα είδους δημόσια υπηρεσία, κοινοφιλή υπηρεσία, ούτε στην αγορά εργασίας. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότιμη μεταχείριση. Οπότε αυτά που είπε ο κύριος Πρόδουερ στην αρχή της παρουσίασής του. Είναι δύσκολο να βρούμε αξιοπρέπεια για αυτούς τους ανθρώπους, τους διάφορους καταβλισμούς. Η Ελένα και εγώ, η συναδελφός μου και εγώ, είναι το εξή. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε κάτι θετικό, μια, μια θετική συνεισφορά. Πολιτική κάνουμε εμείς. Θέλω να υπογραμμίσω ότι για να πετύχουμε το στόχο μας, καταρχήν πρέπει να δούμε τα πράγματα τομεακά. Ενώ να υπάρχει χωριστή μνήα σε διάφορους τομείς. Εκπαίδευση, πρώτα απ' όλα. Αναφέρθηκε από τον κύριο Αμπρόζη το θέμα της εκπαίδευσης. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και πρόσβαση σε άλλες κοινοφιλείς υπηρεσίες. Θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη επίσης για καλή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Και ξέρω για τι πράγμα μιλάω, γιατί σε κάποια άλλη στιγμή τη ζωή μου ήμουνα ε, δημοτική αρχή. Και χρειάστηκε να αναλάβουμε εμείς το βάρος της αλληλεγγύης για άλλη περίπτωση μετατόπισης πληθυσμών. Από την αρχή ανακοίνωση χαρτογραφεί τους πρόσφυγες ανά τον κόσμο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το 86% αυτών ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και 75% οι λιγότερο αναπτυγμένες. Οπότε, ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των χωρών υποδοχή, αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοιες μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμού. Έτσι όπως το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι είναι θετικό. Αναφέρεται στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ε, αναπτυξιακή συνεργασία και προστίθεται, όπως είπε και Ελένα, και η πολιτική διάσταση. Έχω βέβαια κάποιες αφιβολίες ή ερωτήσεις, αλλά είναι αργά τώρα, τέτοια ώρα. Θα απλοποιήσω. Για να δούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την έγκαιρη προειδοποίηση. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά συγκρούσεις μόνο ή έχει να κάνει και με καταστάσεις όπου βρίσκονται διάφορες περιοχές του πλανήτη μας οι γείτονες χώρες που κατά πρώτον θα υποδεχθούν τους πρώτους εκτοπισμένους. Κάποιος από σας χρησιμοποίησε τον όρο μοιραίο για έναν καταβλισμό όπου είπατε ότι θα διαλυθεί. Μα εκεί έχουμε την έγκαιρη προειδοποίηση. Γιατί τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς, αν διαλυθεί ένας καταβλισμός, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε με αυτούς που είναι από το 79 εκεί. Δεύτερον, α, και υπάρχουν εκεί μαζικές μετατοπίσεις εξαιτίας της διπλής κρίσης στο Τσάντ, Μποκοχαραμ και ξηρασία. Απερίμωση. Δεύτερον, τα έγγραφα στα οποία αναφέρεστε στη σελίδα 8 της ανακοίνωσής σας, αναφέρουν μία προληπτική ανάλυση όσον αφορά την προετοιμασία των χωρών εταίρων για να μπορέσουν να υποδεχτούν χιλιάδες ανθρώπους. Μπορούμε να έχουμε κάποια ιδέα, παρακαλώ, για τη δυνατότητα ανταπόκρισης και απορρόφησης. Και τέλος, εκπαίδευση, έτσι. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την εκπαίδευση και δεν ξέρω αν η Επιτροπή είναι σε θέση να μου απαντήσει. Προτείνει η Επιτροπή οικονομική στήριξη και λειτουργική στήριξη για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Τι είδους δηλαδή οικονομική στήριξη σκέφτεστε. Κονδύλια από πού και θα συμπεριληφθούν και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2017. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τόσα μας είπατε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη διαχείριση ροών ή για τον έλεγχο των ροών αυτών, αλλά εγώ από τις δικές μου εμπειρίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σας λέω ότι οι ροές από περιοχές ε, σε πολεμική σύγκρουση σταματούν όταν σταματάει η σύγκρουση. Και μέχρι τότε πρέπει να είμαστε σε θέση να τις διαχειριστούμε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ολόκληρη έκθεση έκανες. Δεν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά με σμάκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Καλωσορίζω και εγώ την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 60 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία εκτοπισμού, κρίση που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις ροές αυτές. Οπότε ναι, ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση, την περιμένουμε εδώ και καιρό Όντως χρειάζεται στήριξη στις περιοχές και να λάβουμε υπόψη μας και τις μελλοντικέ προοπτικές. Αν εγώ ήμουνα στην ε, κατάσταση αυτή που βρίσκονται τώρα οι πρόσφυγες, ήμουνα σε ένα καταβλισμό κάτω από τις συνθήκες που βρίσκονται αυτοί, ίσως και εγώ θα πλήρωνα κάποιον λαθροδιακινητή για να με μεταφέρει εμένα και τα παιδιά μου σε μια καλύτερη ζωή. Άρα χρειάζονται καλύτερες συνθήκες ε, εκπαίδευσης, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ζωτική σημασίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση, να ενισχύσουν δηλαδή τις πρώτες χώρες υποδοχής των προσφύγων για να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Τώρα, για κάτι που είπε η κυρία Χαλτ. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου λίγο πολύ λέει ότι είναι σημαντικό να έχουμε στοιχεία να συγκεντρώσουμε στοιχεία όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση, την αναπτυξιακή κατάσταση και να έχουμε και συγκεκριμένε αναλύσεις για τις ε, μετακινήσεις πληθυσμών, τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών. Είναι ζωτική σημασία εμπειρικά να ξέρουμε τι γίνεται και να οδηγηθούμε στι σωστές πολιτικέ. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι υπάρχει, έχουν συζητήσει για αυτήν την εμπειρική ανάλυση προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Τι μέτρα πολιτικής έχουν οδηγήσει σε κάτι θετικό και ποια όχι. Βέβαια δεν ισχύουν τα ίδια για όλες τις περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς λοιπόν θα κάνει τη διάκριση για να ανταποκριθεί διαφορετικά στην κάθε περιοχή. Και έπειτα η ανησυχία όσον αφορά τις χώρες υποδοχής. Έχετε την αίσθηση ότι πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασία, σε βασικές υπηρεσίες υπάρχουν. Μπορεί να υπάρξει μια μόνιμη κατάσταση με αυτά τα δεδομένα. Μερικές φορές πρέπει να σκεφτούμε ότι τρίτες χώρες μπορεί να μην θέλουν να συνεργαστούν πια μαζί μας. Τι θα κάνουμε. Και έρχομαι τώρα και στην Ουκρανία, που δεν είναι πολύ μακριά από τις χώρες μας. Πρόσφατη κρίση, πριν από δύο χρόνια ακριβώς ανατολικά ε, της Ουκρανίας, είχαμε την πρώτη περίπτωση εσωτερικής ε, τέτοιας ε, μετακίνησης. Με μισό εκατομμύριο, πάνω από μισό εκατομμύριο, είναι οι εσωτερικά μετατοπισμένοι η διεθνής βοήθεια που υποσχέθηκε η διεθνής κοινότητα είτε δεν έχει πάει είτε έχει πάει πάρα πολύ αργά. Έγκαιρα πρέπει να σχεδιάζουμε, ώστε έγκαιρα να σκεφτόμαστε σενάρια για τέτοιες λύσεις. Τώρα δεν το κάναμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σέμποκ. Κυρία Έμποκ, ευχαριστώ πολύ και εμείς ως πράσινοι χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν και θέλω να σας ευχαριστήσω τους ομιλητές γιατί δεν παρουσιάσετε μοναχά τις τεχνικές πτυχές αλλά τονίσατε ότι εδώ πρόκειται για ένα ανθρώπινο θέμα και είναι ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Ακούσαμε σήμερα την Προεδρία της Σλοβακίας ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξης και έχουν τονίσει ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με πολιτικούς που είναι δραστηριοποιημένοι στον τομέα της ανάπτυξης για να αντιμετωπίσουν την, ε, με τις ροές και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μακροχρόνια σχεδιασή και πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το υποστηρίζουμε. Έχω ένα ερώτημα. Για σας είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στις τοπικές οικονομίες οι άνθρωποι αυτοί. Μιλήσατε επίσης και για την ισότητα των φύλων. Ε, αυτό είναι αντιφατικό με αυτό το οποίο ισχύει για την ενσωμάτωση στην αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά. Θα πρέπει να δώσουμε και καλά παραδείγματα για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα. Χωρίς να κατονομάσουμε κάποιες χώρες ή να τις επικρίνουμε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις ε, χώρες αυτές όπου τα πράγματα ίσως είναι καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τσέρερ, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πρότασή της. Για μένα όμως, όλα από αυτά τα πράγματα που αναφέρονται είναι για μένα σχεδόν προφανή αναφέρεται ότι πρέπει οι πολιτικοί και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται για τα θέματα ανάπτυξης συγχρόνως θα πρέπει να συνεργαστούν και με αυτούς που αντιμετωπίζουν τα θέματα της ε, ανθρωπιστικής κρίσης από τη στιγμή που ξεκινάει μια κρίση. Εμείς έχουμε δει στην ε, δεκαετία του 1990 πολύ μεγάλα προβλήματα όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την πρώην Ιουκοσλαβία. Γιατί όμως δεν κάναμε κάτι τέτοιο ενώ όλοι το θεωρούμε προφανές. Λυτούμε από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν. Αλλά γιατί δεν έχουν δράσει με τον τρόπο αυτό και λέμε μετά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ποιον εννοούμε. Έχουμε μια ένωση κρατών μελών που πρέπει το καθένα από αυτά τα κράτη-μέλη να αναλάβει την ευθύνη αυτή, να την επομιστεί. Αλλά βλέπουμε ότι ο καθένα την κάνει πάσα στου άλλου την ευθύνη αυτή. Πώ θα εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει με ενωμένο τρόπο για τα θέματα αυτά και είδαμε πρόσφατα ότι ακόμα και με το θέμα της εσωτερικής μετακίνησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ελεύθερης μεταδιακίνησης έχει υπάρξει μια εκστρατεία η οποία βασίστηκε σε αυτό ακριβώ το θέμα για να ζητήσει και να επιτύχει την έξοδο μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο εάν το θέλουμε. Στην πράξη δηλαδή πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα και όχι να παραμείνουμε μονάχα στη σφαίρα της θεωρίας. Και επομένως να ασκήσουμε και πίεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή στο Νότιο Σουντάν βλέπουμε ότι δεν μπορούν και αυτοί που έχουν την εξουσία να ελέγξουν τα στατεύματά τους και δεν μπορούν να εμποδίσουν τον κόσμο εκεί να πυροβολείται μεταξύ του και παρά τις εκκλήσεις για ειρήνη και ομαλότητα δεν γίνεται τίποτα και εξακολουθούν οι μάχες εκεί. Επομένως κατανοώ την ε, έκκλησή σας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια και των κρατών μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν στην πράξη με ενιαίο τρόπο ώστε να μην μπορεί ο καθένας να κρύβεται πίσω από τον άλλο και να μεταθέτει τα προβλήματα αλλού και να δημιουργούν καταστάσεις ανασφάλειας του πληθυσμού και το οποίο οδηγεί και σε μεγάλο, μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Στην Γερμανία, παραδείγματος χάρη, για την ενσωμάτωση των μεταναστών ε, χρειάστηκε να δαπανηθούν 25 δισεκατομμύρια στον προηγούμενο χρόνο και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα χρειαστούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά για να υπάρξει πρόσβαση στην αγορά των ε, μεταναστών. Αυτό προϋποθέτει γνώση της γλώσσας μιας χώρας και να υπάρξει και μια προσαρμογή του προφίλ δεξιοτήτων των ανθρώπων αυτών προς την αγορά εργασίας και όλα αυτά φυσικά κοστίζουν να υπάρξει αυτή η κατάρτιση και η γλωσσική μάθηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να υπάρξει ένα αξιόπιστο πλαίσιο, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διακρίνω να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώ. λέει ο πρόεδρο. πιεζόμαστε πάρα πολύ από το χρόνο. Έχουμε το πρόβλημα με του διερμηνεί. Μπορώ να σα δώσω με το ζόρι τρία λεπτά σε έκαστον των τριών. Προσπαθήστε να απαντήσετε στα όσα σα ερώτησαν. Ο κύριο Γενικό Διευθυντή. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Ντεμπρούγερ. Είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε με τέτοιο συνοπτικό τρόπο. Κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία αναφέρθηκαν στις διάφορες παρεμβάσεις. Η εταιρική σχέση και ο διάλογος με τις αρχές των χωρών της προέλευσης, των χωρών υποδοχής και με τις τοπικές αρχές. Αυτά είναι στοιχεία κλειδί για την νέα αυτή πολιτική, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποιους τέτοιους συνομιλητές πρώτα απ' όλα. Αναφέρθηκε το στάδιο του αν βγει από αυτή την κρίση. Αυτό θα μπορέσει να γίνει μονάχα με ένα ανοιχτό διάλογο με την κυβέρνηση της Κένιας και της Σομαλίας, με τις τοπικές αρχές της Σομαλία και με άλλες χώρες και οργανώσεις περιοχής. Παραγωγής χάρη σκέφτομαι στην Αιθιοπία ή την Ουγγάντα. Θα πρέπει όλες αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν στην επίτευξη μιας λύσης για αυτή την κρίση η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Αυτό αναφέρθηκε από ορισμένου συνεισηγητές. Μιλήσαμε για την υγειονομική περίθαλψη, την παιδεία, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τις δημόσιες υπηρεσίες εν, εν γέν. Αλλά εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα γιατί αυτή η πρόσβαση δεν μπορεί να γίνει με ανταγωνισμό των τοπικών ε, των Ιθαγενών πολιτών και των ανθρώπων που έρχονται ως μετανάστες ή πρόσφυγες. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισότιμη μεταχείριση και εκεί θα διακυβευτεί η, επίτευξη, η επιτυχία ή η αποτυχία ενός προγράμματος αναπτυξιακού χαρακτήρα για τα άτομα αυτά σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Οι υπηρεσίε που αναφέραμε ως προηγουμένως είναι απαραίτητες. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση όλων αυτών των εργασίων είναι στον τομέα της παιδείας. Προσπαθούμε να το κάνουμε στο Λίβανο, προσπαθούμε να το κάνουμε στην Τουρκία. Θα το κάνουμε και στην Ελλάδα στο μέλλον. Πρόκειται για μια εδραίωση του συστήματος παιδείας επιτόπου στις χώρες υποδοχής για να μπορέσουν να απορροφήσουν τους νέους αυτούς φοιτητές και μαθητές από τους μετακινηθέντες. <clears throat> Αλλά συγχρόνως αυτή η εδραίωση των αισθητικών συστημάτων θα πρέπει να ενισχυθεί με μια προσπάθεια σε έκτακτη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι η προτεραιότητα του Επιτρόπου στη Λιανίδη, ώστε να μπορέσουν και οι ανθρωπιστικοί φορείς να προετοιμάσουν αυτά τα παιδιά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέους ε, χώρους εκπαίδευσης. Για την ανάλυση των αναγκών και τις έγκαιρες προειδοποίησης θα έλεγα στον κύριο Διάς ότι η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η δεύτερη έννοια που πρέπει να αναφέρουμε δεν έχει να κάνει μονάχα με την ανάλυση των συγκρούσεων, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά και την τεχνική ανάλυση των αναγκών, τόσο και για τα άτομα τα οποία εκτοπίζονται και για τις κοινότητες υποδοχής. Αυτή είναι μια δέσμευση όπου πρέπει να εμπλακούν οι δωρητές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως έκαναν στην Παγκόσμια ε, Ανθρωπιστική ε, διάσκεψη και με την προσέγγιση που ακολούθησε η κυρία Γιώργεβα που είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Επειδή τέθηκε το θέμα της Ουκρανίας, είμαστε όλοι ιδιαίτερα ε, προσεκτικοί για την κατάσταση της χώρας αυτής. Εκεί έχουμε εστιάσει την ανθρωπιστική βοήθεια εκεί που υπήρχε πραγματική ανάγκη, δηλαδή στις εμπόλεμες ζώνες είναι τεράστιο το βάρος των εκτοπισμένων ατόμων, αλλά ξέρουμε ότι είναι και η πρώτη ευθύνη της Ουκρανικής κυβέρνησης πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αμπρόζη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Μια που δεν έχουμε χρόνο, έχω δύο παρατηρήσεις. Για όσα είπε ο Λουί, πρώτα πρώτα παρατήρηση, μας ανέφερε το ζήτημα αυτών των πρόσφατων μετακινήσεων προς Ευρώπη και το ζήτημα της ασφάλειας αλλά και του ελέγχου των ροών για λόγους ασφαλείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι το οποίο ίσως δεν είναι και τόσο προσφυλές στον κόσμο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι δηλαδή βάσει της ε, εμπειρίας μας, εμπειρίας δεκαετιών, ξέρουμε ότι όσο πιο κατασταλτικά είναι τα συστήματα για την πρόσβαση, για μετανάστευση, για πρόσφυγες, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ροή. Οπότε αυτό ισχύει και για συνοριακούς ελέγχου ισχύει για κατασταλτικά περιοριστικά μέτρα για τη μετανάστευση, αλλά για την πρόσβαση των προσφύγων εκεί που ψάχνουν προστασία. Οπότε και έτσι επίσης αυξάνουμε και την γκρίζα ζώνη της παράνομης ε, διακίνησης. Άρα δεν υπάρχει ο έλεγχος και άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση και καλύτερο έλεγχο μεγάλων ροών προσώπων θα πρέπει να έχουμε επαρκή νομικό μηχανισμό και για την ε, προστασία και για την πρόσβαση όλων των μεταναστών και προσφύγων που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αλλού ισχύει αυτό που σας λέω. Νομικό πλαίσιο όχι μόνο για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες. Έχει βελτιωθεί αυτό αλλού στον κόσμο και αυτό πολλές φορές ωφελεί, ωφελεί και την ασφάλεια. Άρα δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω. Είναι εφαρμογή των όσων ισχύουν αλλού. Τώρα. Έχω άλλες δύο παρατηρήσεις. Αναφέρθηκε το ότι εάν έχουμε διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά απασχόλησης, τι θα γίνει. Μα και αυτό είναι ένας μύθος που θα πρέπει να καταρριφθεί. Διότι ίσως έχουμε κάποιες λίγες περιπτώσεις κάποιον μπορεί να τους ελκύσει η βοήθεια στην Ευρώπη ή κάπου αλλού, θα πρέπει να μην ξεχνούμε επιτέλους το ότι υπάρχει και το αντίθετο. Ότι δηλαδή τα αντικίνητρα ακριβώς με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας θα αυξηθούν αυτά τα αντικίνητρα, λέγω. Δεν έρχονται εδώ γιατί θέλουν να βρουν δουλειά στην αγορά εργασία μας έρχονται γιατί θέλουν να γλιτώσουν από τις βόμβες ή θέλουν να γλιτώσουν από φτώχεια, από πείνα, από απερίμωση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό μετακινούνται. Όχι επειδή θεωρούν ότι εδώ πέρα θα υπάρξει κάποια αρρωγή τους οποιοδήποτε είδους. Άρα επομένως αυτού του είδους η μεταβλητή του κινήτρου να ληφθεί υπόψη ληφθεί υπόψη σημασία. Τώρα, τελευταία παρατήρηση. Μα είπατε για την έγκυρη προειδοποίηση κλπ. Και για το κατά πόσον η διεθνή κοινότητα προβληματίζεται για το τι να κάνει. Αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της επιστροφής στην Σομαλία ε, σημαντικού αριθμού ανθρώπων. Τι συνέπειε θα έχει στη χώρα αυτή η μαζική επιστροφή, αλλά αυτό ισχύει και για τι ευρωπαϊκέ πολιτικές. Να σκεφτούμε δηλαδή τι αποφάσεις έχουν ληφθεί, τι προγράμματα έχουν τρέξει για όλες αυτές τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές και βασικός άξονας της δράσης στην Ένωση είναι η επιστροφή Λέμε να αυξηθεί η επιστροφή, να αυξηθεί ο ρυθμός επιστροφής, να, να γυρίσουν αυτοί που δεν έχουν νόμιμο λόγο παραμονής. Εντάξει, είναι σημαντικός μηχανισμός η επιστροφή, αλλά ας κάτσουμε να σκεφτούμε πώς και τι κλίμακας επιστροφή θέλουμε. Γιατί δεν είναι το ίδιο να επιστρέψουν 10.000 στην Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία ε, και το να γυρίσουν 10.000 στο Μογκαντήσου δεν είναι ίδιες οι επιπτώσεις και οι συνέπειες. Οπότε εντάξει για να προετοιμαστούμε για το μέλλον σύμφωνοι και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων μας να κάτσουμε να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειες αν το κάνουμε ή αν δεν το κάνουμε. Οπότε μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η ιδέα είναι καλή αλλά αν δεν εφαρμοστεί σωστά θα τα κάνει χειρότερα. Ε, ευχαριστούμε. Για ναι πάρα πολύ σύντομα. Ελέγχθηκαν πολλά από τους συναδέλφους μου. Για τον κύριο Ντεμές Μάκερ. Θέλω να σας πω ότι, ότι πράγματι έχουμε πολλά παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι κοινότητες υποδοχής και οι άνθρωποι που είναι εκτοπισμένοι είχαν μια ευτυχισμένη συμβίωση και η ενσωμάτωση ήταν επιτυχής, αλλά δεν συμβαίνει αυτό πάντα και χρειάζεται πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν και η συμμετοχή των τοπικών αρχών και είναι και θέμα πόρων, ώστε οι δύο κοινότητες να μην θεωρήσουν η μία την άλλη ως ανταγωνιστές για τους ίδιους πόρους, αλλά να καταλάβουν ότι όλοι εποφελούνται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες για να το κάνουμε αυτό και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στις προτάσεις για λύσεις και αυτή η προτινόμενη πλατφόρμα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για την επόμενη ομιλήτρια για αυτά που είπε για την ανάγκη να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας οι άνθρωποι αυτοί που μετακινούνται και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ομοσπονδία Κρατών πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Δεν πρέπει να σπρώξουμε στις γειτονικέ χώρες όλη την ευθύνη για χώρες όπως η Τουρκία ή η Ορδανία που υποδέχονται εκατομμύρια πρόσφυγων, πάνω από τρία εκατομμύρια στην Τουρκία και τους ζητούμε να ανοίξουν και την αγορά εργασία σε αυτούς τους ανθρώπους όταν στη Δανία έχουμε 8.000 πρέπει να υπάρχει και κάποια έννοια αναλογίας και μέτρου σε όλα αυτά, αλλιώ δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα με τις χώρες αυτές. Μετανάστες από τη Συρία, όπως είπε η κυρία Βαλενσιάνο, για τους λίγους που έχουν καταγραφεί. Εγώ ήμουν τότε στον Ερυθρό Σταυρό και επικεφαλής της ε, ανταπόκρισης που δόθηκε στους ε, μετανάστες το 2012 και στην αρχή και στην Ιορδανία και στον Λίβανο τους υποδέχτηκαν σαν αδέλφια, σαν φίλους και επισκέπτες πάρα πολύ δεν καταγράφηκαν γιατί δεν περίμεναν θα μείνουν στην προσφυγή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν λοιπόν <clears throat> ιστορικοί λόγοι γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν ήδη στην Ιορδανία, είχαν κατασταθεί, είχαν τις επιχειρήσεις τους που έχουν φτιάξει εκεί, όλα αυτά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα και λεπτά θέματα. Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι μου έχουν πει ήδη πολλά. Ευχαριστούμε τους ειδικού και ευχαριστούμε και την Επιτροπή ΔΕΒΕ που ήρθε να συμμετάσχουν εδώ με την ΑΦΕΤ. Στις 29 Αυγούστου θα είναι η επόμενη συνάντησή μας. Καλό βράδυ και καλές διακοπές. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς.